Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών μας, του ελέγχου του προϋπολογισμού και προϋπολογισμών. Θα... Ε, ήμουν πανευτυχής μπορούσα να δώσω το λόγο στην Ίγκε Γκρέσλε, η οποία με μεγάλο κύρος και μεγάλη πραγματογνωμοσύνη διεξήγαγε τις πάρα πολλές ε, συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου που κατέληξαν σε συμφωνία με το Συμβούλιο για το σχέδιο αναθεώρησης και απλούστευσης του δημοσιονομικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η κυρία Γκρέσλε κολλείεται λόγω προβλημάτων μεταφορών και δεν θα παραστεί στην σημερινή συνεδρίαση. Θα παρακαλέσω τον συνεισηγητή μας, τον Ρίτσαρτ Άσουορθ, να μας πει τα βασικότερα σημεία ε, πριν ψηφίσουμε το κείμενο στο σύνολό του. Θυμίζω ότι πρόκειται για μία ψηφοφορία ενιαία που αφορά τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο με στόχο να καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση σε συμφωνία για την προστασία τροποποίησης του λόγω δημοσιονομικού κανονισμού. Το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας ε, δέχτη τις ευλογίες του Κορυπέρ την περασμένη Πέμπτη και έχει και συμβουλευτική επιστολή του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου φυσικά θα περάσει και από τους νομομαθείς ε, και γλωσσομαθείς νομικούς ε, πριν φτάσει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Και στην Ολομέλεια θα εψυναυθούν πολιτικές ε, δηλώσεις. Ελπίζω τα αποτελέσματα να είναι στο των φιλοδοξιών μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απλούστευση, για να μην μας υποφτευτεί κανείς για παραπλανητική διαφήμιση κανείς από τους δικαιούχους ε, των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Μόνο στην πράξη ε, θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στον κύριο Ashworth που είναι συνεισηγητής εκτός από την κυρία Γκρέσλε. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι εδώ στην ψηφοφορία για την ψήφιση της εκθέσεως. Όπως ερχόμουν σκέφτηκα ότι ίσως αυτό είναι ρεκόρ του Κοινοβουλίου. Είναι η πιο μακροσκελής έκθεση και πιο σύντομη ψηφοφορία. 700 σελίδες περίπου είχαμε κειμένο που επεξεργαστήκαμε. Και ήμασταν μαζί Πρόεδρε, είχαμε περίπου 40 τριμερείς τριλόγους. Ε, ο κάθε διάλογος κάτι σε τουλάχιστον ένα τρίωρο. Και να καταλήξουν σε ψηφοφορία είναι τα κρονάτων της απλούστευσης. Απλούστευση. Hm. Είναι ο μύτος Αριάδνης. Είναι το νήμο που διασυνδέει τις προσπάθειες για το δημοσιονομικό κανονισμό. Απλούστευση τι σημαίνει Θέλουμε η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να είναι ευχερέστερη. Θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό εξετάσαμε όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες. Συνάδελφοι, οι ελεγκτικές διαδικασίες, και είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να είναι στεναρές, ισχυρές, να αποφύγουμε τις απάτες και τις καταχρήσεις. Όμως, ένα από τα προβλήματα που είδα είναι ότι στην επιδίωξη της απλούστευσης ανεφάνει κι άλλος στόχος. Ο υπολογισμός σου κατατίζεται βάσει επιδόσεων. Εσόμενοι στραφής βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση του υπολογισμού θα μειώνεται ενώ οι απαιτήσει από τον υπολογισμό θα αυξάνονται. Έτσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι Ευρωβουλευτές θα πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις τους και τι προτεραιότητες τους συναρτήσει της κατανομής των πόρων βάσει στοιχείων ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για τα χρήματά μας. Άρα κατάτηση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων. Είναι πρώτες ημέρες αυτής της προσεγγίσεως. Στο μέλλον θα ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες και θα είμαστε αποτελεσματικότεροι. Όμως ήθελα να το υπογραμμίσω, διότι είναι σημαντικό στοιχείο. Κάποια παραδείγματα αυτών που κάναμε για την απλουστευμένη διαδικασία και την υποβολή αιτήσεως για διοικητικές χορηγίες. Και οι πληρωμές συναρτώνται με τα αποτελέσματα. Σαφήνεια επικρατή, αναλογικότητα και σωστά ελεγκτικά συστήματα. Η θέση του Κοινοβουλίου ενισχύθηκε παρέμειναν οι αρμοδιότητες όσον αφορά τα θέματα του προπολογισμού. Και η κατανομή των χορηγιών σχετίζεται με την μη ε, κερδοσκοπία. Εξετάσαμε νέα μέσα, όπως το καταπιστεύματα. Υπενθυμίζω εδώ ότι απορρίψαμε τη χρήση των καταπιστευμάτων για εσωτερική διαχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει τα νέα εργαλεία τα οποία εμείς δημιουργήσαμε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Συζητήσαμε το αποθεματικό για κρίσεις. Επίμαχο ζήτημα. Λύθηκε το πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικές Επενδύσεις για το ΕΦΣΙ. Και τι σχέση έχει αυτό με τη συμβατική χρηματοδότηση μέσω της κατηγορίας 1 του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τέλος, άλλο εμπόδιο ήταν η ημερομηνία εφαρμογής. Κανονικό θα ήταν να θεσπιστούν νέοι δημοσιονομικοί κανονισμοί που θα αρχίσουν από πρώτη πρώτου. Όμως, οι άλλες ε, επιτροπές μέσω των διαδικασιών διαπραγματεύσεων όμνιμους έχουν άλλες πρακτικές, όπως η Επιτροπή η Περιφερειακή και για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Γίνεται καταστρώματα εφαρμογή και είναι αποτελεσματική προσέγγιση. Έγινε πολλή δουλειά, όπως σας είπα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες ευχαριστίες τώρα. Πρώτα απ' όλα απευθυνόμενος προς το Συμβούλιο, που δεν είναι παρόν, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι η Εστονική Προεδρία, κυρίως μας της Σάιερ, που έκανε 99% εκπροσωπός της, της δουλειάς, πολύ καλή δουλειά, αποτελεσματικότατη, εντυπωσιάστηκα από αυτά που έκαναν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Νάντια Καλβίνο και η ομάδα της έκαναν προσπάθειες. Τους ευχαριστώ. Και τον Επίτροπο, τον κύριο Έτιγκερ, να μην τον λησμονούμε. Τέλος. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές. Τους ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία τους. Από την αρχή της προσπαθίας. Έκανε τεράστιες προσπάθειες. Ευχαριστώ και εσάς, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, για την υποστήριξή σας για τις συνετές σας συμβουλές. Τις εξετίμησα ιδιαίτερος. Προσπαθήσατε και πέρα από τα πλαίσια των καθηκόντων σας. Και σας ευχαριστώ και το αναγνωρίζω αυτό, όπως και άλλοι εισηγητές. Ευχαριστώ και την Inge Κρέσλε. Χωρίς εκείνη δεν θα τα καταφέρναμε. Είναι ατυχές που δεν παρήσατε σήμερα. Η Inge ζει και αναπνέει δημοσιονομικό κανονισμό. Εκ μέρους του Προέδρου, του κ. Αρτουή, και εκ μέρου μου που είμαι συνεισηγητή πρέπει να πω μα διευκόλυνε τη ζωή. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα χωρί την γκια και την ομάδα τη. Έκαναν υπέροχη δουλειά. Εκφράζω τι ευχαριστίε μου απευθυνόμενο προ αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με όλες τις ευχαριστίες και να προσθέσω και το όνομα του Ρίτσαρτ Ashworth και ας τους χειροκροτήσουμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη τόσο σημαντική δουλειά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των διαδικασιών, εγώ είχα ζητήσει να υπάρξει μεγαλύτερη απλούσταυση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι εκτελούμε τώρα ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μέχρι εκεί δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα από όσα ήδη επιτύχαμε. Αλλά δεδομένων όλων αυτών των συνδικών, γιατί προετοιμάζουμε τώρα και το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν θα ήθελα να μου πούνε ότι εντάξει τώρα τα αποφασίσαμε και αυτή την απλούστευση που αποφασίσαμε στην προηγούμενη περίοδο θα την εφαρμόσουμε και τώρα και θα, μεταφερθεί μετά το 2014-2020. Απευθύνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2020-2027 να έχουμε νέα απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού, διότι αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ συχνά και όχι, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν ε, όλα αυτά που τους επιβάλλουμε, γιατί χωράει και ακόμα περισσότερη απλούστευση, πιστεύω. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να ρυθμίσουμε το sponsoring και ο καθένας αναρωτιόταν τι είναι sponsoring. Και είπαμε, ή μας είπαν μάλλον, ότι θα πρέπει να είναι σε μετρητά. Α, ε, όχι, μάλλον να μην είναι σε μετρητά, σε είδος για τους εκπροσώπους μας στις διάφορες αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, τους πρέσβεις που υπηρετούν εκεί και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, την 9η Μαΐου. Και συχνά δεν έχουν χρήματα για να διοργανώσουν εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, δεξιώσεις, σαμπάνια, καναπεδάκια κτλ. Να δεχθούν τον κόσμο. Και αυτό είναι το sponsoring. Χορηγία, όχι σε χρήμα, αλλά σε είδος, τα καναπεδάκια. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας κάνουμε λοιπόν μια δοκιμαστική. Η ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Est-ce que tout le monde a voté Non. Ψηφίσατε όλοι. Έχω 25 εγώ που ψηφίζουν. Voilà, tout Πέρας. Κάποιος δεν έχει κάρτα. Την ξεχάσατε στο Στρασβούργο στο μηχάνημα. Ωραία. διανατάσει ο σχηρός. À Ψηφίζουμε λοιπόν όλο το κείμενο όπω προέκυψε από τη συμφωνία στον τριμερή διάλογο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ενημερώνουμε στην κλίση βεβαίως. Scrutin Λοιπόν, εσείς τι ψηφίζετε, συνάδελφε, που δεν έχετε την κάρτα σας. Υπέρ ψηφίζετε. Αποχή. Αποχή, αποχή. Λοιπόν, 21 υπέρ, 1 Κατά και τέσσερις αποχέ, λέει ο πρόεδρος. Όχι, αποχή είπε ο κύριο που δεν έχει την κάρτα του. Α, πέντε λοιπόν και είκοσι υπέρ. Εγκρίνεται το κείμενο. Υπερψηφίζεται. Ωραία, εξαντλήσαμε και την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τη συμμετοχή σα. Και συγχαρητήρια στου δύο συνεισηγητέ. Richard Ashworth et